με την κατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Κασκάρ, Σινγκιάνγκ, αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων στην Κίνα. Και καταρχήν θα δώσω λόγο στους συντάκτες και πρώτα στον κύριο Κέλαμ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. η γόροι είναι μία ε, μειονότητα στην ε, ιστορική κοιτίδα τους και πρέπει να μπορέσουν να διατηρήσουν ότι ε, ταυτότητά τους. Το πρόγραμμα εξυγχρονισμού έχει ζητήσει να καταστραφεί σταδιακά το Κασκάρ, αρχαία πόλη του δρόμου του μεταξιού και εάν οι κινέζικες αρχές ε, είναι σοβαρές ε, θα πρέπει να, να μπορέσουν να πείσουν τουλάχιστον τους αυτόχθονες ότι θα προστατευθεί η πολιτισμική τους κληρονομιά και θα μπορέσουν να μην ισοπεδωθούν από τα κινέζικα ήθη και Υπάρχει μία πολύ σημαντική ε, εμπειρία στο θέμα της προστασίας Τη της πολιτιστικής και ζητώ από τους Κινέζους να διατηρήσουν ορισμένα πολιτιστικά κοιμήλια στο δρόμο του μεταχιού. Τώρα η κυρία Σάκη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Επίτροπε, συνάδελφε, για το θέμα ε, μάλλον στο όνομα της ε, εξέλιξης και της προόδου καταστρέφεται η αρχαία πόλη του Κασικάρ. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλάπτει την πολυμορφία, την πολιτιστική της Κίνας που, που καταστρέφεται. Η Κίνα θέλει να προωθήσει τις την πολιτιστική διπλωματία. Κανείς όμω δεν θα ενδιαφέρεται για μια εξυγχρονισμένη χώρα η οποία καταστρέφει την πολιτιστική της ε, ε, κληρονομιά. Βιώσιμε σχέσεις με το υπόλοιπο κόσμο, ε, σεβασμός ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικός γι' αυτό. Εμείς καλούμε την κινέζικη κυβέρνηση να εκτιμήσει το ενδεχόμενο σε μια κοινή αίτηση με το Καζακστάν, το Κυργιζιστάν και το Σμπεκιστάν να ζητήσουν να ε, αναγνωριστεί ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά των Ηνωμένων Εθνών ε, το Κασγκάρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Σάκ και δίνω το λόγο στην κυρία Γκέρι Ντεότεμπερ για ένα λεπτό. Το ζήτημα αυτό το, ε, το εξετάζουμε μετά από την, ε, όσα μάθαμε από τον Ταρελάμα για την απελευθέρωση κάποιων ε, κάποιους κρατούμενους. Τώρα μιλάμε για μια άλλη μειονότητα, αυτή των ε, Ουιγούρων στο Σιάνγκ. Η Κίνα διολογεί τη στάση της με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να καταστρέψει την πολιτική κληρονομιά. Το θέμα της σταδιακής ε, καταστροφής του Κασκάρου νομίζουμε ότι είναι μια πράξη η οποία θα πλήξει ιδιαίτερα την ε, πολυσυγκρονομία της περιοχής. Κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες ε, μεταβαίνουν στην περιοχή παρακαλώ να ζητήσουμε από τις διευρωπαϊκές αρχές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να καταστούν πιο αποτελεσματικές και στις συζητήσει που θα έχουν με την Κίνα να θίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι μειονότητε αλλά και το ζήτημα της πολιτική Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία ε, ε, Έτεμπερ και ακολουθεί η κυρία Μπράπελς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Κασκάρ είναι το σύμβολο κατά τεξοχήν της ε, περιοχής του ε, Ανατολικού Τυρκιστάν ε, και είναι στα σύνορα της Κίνας. Είχα διοργανώσει μία συνεδρίαση και είδα τις επιπτώσεις της καταστροφής αυτής επί του λαού διότι υποτίθεται ότι υπάρχει ε, εξασφάλιση αλλά ε, δεν πρόκειται να μείνει ούτε ο μισός πληθυσμός οπότε πρέπει να προχωρήσουμε πριν να είναι πολύ αργά διότι ο λαός αυτός κατακρίνει την ε, κυβέρνηση διότι ε, τέστηλε τις άλλες εξεγέρσεις ή στο παρελθόν και θα πρέπει να υπάρξει μία απονομική πολιτική στην περιοχή κατά τρόπον ώστε να προστατευτούν αυτά τα πολιτιστικά αγαθά της ε, κληρονομιάς των Ουιγούρων αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε κινήσεις μπορεί να γίνουν κατά το, της των κατοίκων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι σε αυτές θα θεωρηθούν μια ε, πολιτιστική ε, των μειονοτήτων. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφο. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, ένα τέτοιο συνέστημα σαν αυτό που συνήθως ακούμε δεν υπάρχει στην Κίνα και δεν σκέφτεται κανείς να εορτάσει την ε, διαφοροποίηση αντιθέτως ε, σε μια πολυπληθή χώρα καταστρέφεται η κληρονομιά των μειονοτήτων πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλη δυστημία όπως άλλο είχε ήδη γίνει για το Θιβέτ και τώρα γίνεται για το Κασκάρ που ήταν μια εξέχουσα πόλη στο δρόμο του μεταξιού και τώρα πρέπει να καταστραφεί και να ανοικοδομηθεί. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί το Πεκίνο να ε, καταστήλει το πνεύμα των ε, ε, Ουιγούρων που θέλουν να αποσχέσουν αλλά μία καταστροφή μιας πόλης σαν το Κασκάρ απλούστατα θα συσπυρώσει όλους αυτούς οι οποίοι θα υποκινήσουν βία κατά του κράτους. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σταβάρης για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για να σας πω την αλήθεια, ανάμεσα στις τρεις συζητήσεις ε, κατεπήγοντα χαρακτήρα που συζητάμε απόψε, ε, αυτή είναι αυτή που εμείς ε, θεωρούμε πιο σημαντική. Μιλήσαμε για το Πακιστάν, για τη Λευκορωσία και να σκεφτούμε όχι μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηθική, ηθικό κύρος, αλλά μπορεί να πιέσει τις αρχές ε, για να μπουν στο σωστό δρόμο. Όμως όταν μιλάμε για την Κίνα, αυτό το πλανέκτημα περιορίζεται πάρα πολύ. Γιατί αυτό είναι αντίθετο με αυτά που κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στις δικές μας πρωτεύουσες. Τα όσα κάνει ο κ. Σαρκοζή, η κυρία Μέρκελ και στη χώρα μου ο κ. Σόκρατες που πολύ πρόσφατα έκανε μια αναδιαδήλωση ε, που ήταν κατά των κινέζικων αρχών να παρακάμψει το χώρο που διέμενε ο Κινέζος ε, αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Οι Κινέζοι έχουν μεγάλη ε, φαντασία, φαντασία και μπορούν να, να λειτουργήσουν, αλλά ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης σε όλες τις ζώνες, είτε είναι Πεκίνο, Σανγκάι ή το Θιβέτε. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο το Ευρωκοινοβούλιο να πει αυτά που θέλει να πει σήμερα και που τα έχουμε γράψει εδώ στο ψήφισμά μας που λέει ζητούμε από τις, κινεζικέ από τις Κινέζικες Αρχές να σταματήσουν αυτή τη δημογραφική δολοφονία ε, και εθνοκάθαρση που κάνουν κατά των Ουιγούρων γιατί μιλάμε για χώρους μεγάλης κληρονομιάς ε, παγκόσμιας κληρονομιάς όμως τελικά ε, οι δικοί μας ηθήνοντες σιωπούν όταν βρίσκονται ενώπιον των Κινέζων ηθινόντων. του τους δίνουν λευκή, λευκή επιταγή αυτό είναι εξελίξεις που τελικά μας κάνουν να φαινόμαστε σαν ε, απλώς να θαυμάζουμε και να απορούμε. Το κύριο μας λοιπόν είναι εδώ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ξαναεπανεξετάσουμε λοιπόν τη στάση μας απέναντι στην Κίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ταβάρες. Τώρα είναι οι ομιλητές εν ονόμα των πολιτικών μηνωμάτων και καταρχήν ο κύριος Πόσελτ για ένα λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, οι Ουγγούροι δεν είναι μειονότητα αλλά ένας πληθυσμό στο δρόμο του μεταχιού από την αρχαιότητα και οι ε, Ουγγούροι ε, έχουν την προστασία του Διεθνούς Συμβουλίου από το Μόναχο και της ομάδος Blue Shield που μας επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα στο Στασβούργο. Οπότε κάνουμε μία φιλική έκκληση προς τους Κινέζους οι οποίοι απειλούν τους Ιουγούρους με μία εθνοκτονία. Θα έπρεπε λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι ε, ένα από τα χαρακτηριστικά ενός πολιτισμού είναι να προστατεύει τους άλλους πολιτισμούς ιδίως όταν είναι μικρότεροι σε ένα γιγαντιαίο κράτος. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη μας ότι ε, σε τρία σημεία λέμε ότι η, κληρονομική, ε, η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιουηγόρων. Και τώρα η κυρία Κρετού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πιστεύω πως ε, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα από όλες τις ε, πλευρές. Δεν ε, χρειάζεται να σκεφτούμε μόνο το θέμα της σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Mm. Η επαρχία του Σιν Γιάνγκ είναι μια απόδειξη προσφυγή στην βία. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τον διεθνωτικό διάλογο. Το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να αναφερθεί στο δυνατότητα και το δικαίωμα της Κίνας να ε, ε, υποστηρίξει κάποιες επαρχίες ή όχι. Το ζήτημα είναι να προσπαθήσουμε εδώ να υποστηρίξουμε τον ε, επαρχίες σε οικονομικό επίπεδο. Ευχαριστώ η κυρία τον επαρχιες σε οικονομικο επιπεδο ευχαριστω η κυρια για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ. η επαρχία των Ιγούρων ε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα δεύτερο Θιβέτ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ε, τη στάση που κρατάει η Κίνα. Ίσως ε, ενδεχόμενα να έχει κατά βάθο στο μυαλό της να καταστρέψει αυτήν την περιοχή. Εμείς όμως δεν πρόκειται να... Δεν πρέπει μάλλον να τους αφήσουμε να καταδαφίσουν το 85% των κτηρίων της ε, παλιάς πόλης ε, του Κασκάρ. Ε, μην ξεχνάμε ότι οι πληθυσμοί ανήκουν σε σκεφτικές μειονότητες. όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σεβαστά από την Κίνα, όπως γίνονται σεβαστά από όλα τα πολιτισμένα κράτη. Η Κίνα επανειλημμένα έχει προθέσει να αποξενώσει κάποιες μειονότητες. Ε, πρόκειται για ε, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε να συμβαίνει τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ την κυρία Ούγιουλαντ. Ακολουθεί ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο οι Κινέζοι φαίνεται να δυσαρεστούνται όταν αναφέρονται άλλοι σημαντικοί πολιτισμοί, ιδιαίτερα τα ιστορικά ε, μνημεία ε, βλέπουμε ότι το Κασγκάρ είναι ένα, από, είναι ένα μνημείο της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων που ζουν εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Γι' αυτό και η κινέζικη διοίκηση προσπαθεί να καταστρέψει τις ε, μικρότερες εκδηλώσεις ε, ταυτότητας, εθνική, εθνικής ταυτότητας και την πολιτιστική κληρονομιά των διαφόρων λαών. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο οι Κινέζοι μπορούν να υιοθετήσουν μια τέτοια, μια τέτοια φιλοσοφία αποδοχής γιατί η σύγχρονη ιστορία τους βασίζεται στη δική τους παράδοση και στην παράδοση ε, αποκλειστικά την Κινέζικη. Η προσέγγιση της Κίνας στο Κασγκάρα αποδεικνύει ότι η Κινέζικη διοίκηση δεν μπορεί να σεβαστεί τη συμβολή άλλων πολιτισμών και εθνών στην ιστορία τους. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι αυτό το σεβόμαστε για να το σεβαστούν και οι Κινέζοι. Ευχαριστώ κύριε Πάσχα, με συγχωρείτε γιατί σας προειδοποίησα πολύ νωρίς. Τώρα υπάρχουν ακόμη ομιλητές και πρώτο κύριο κύριος για ένα λεπτό. Το Κάσκαρ είναι μια πόλη 3,5 εκατομμυρίων ατόμων, δηλαδή λίγο λιγότερο από το συνολικό πληθυσμό της Ιρλανδίας και είναι ε, ένα από τα βασικά σημεία εις το δρόμο του μεταξιού και έχει ε, προστατεύσει την Ισλαμική παράδοση στα πρόθυρα της ε, ερήμου και βεβαίως είναι ένα πολιτισμικό θησαυρός και επειδή όμως οι Κινέζοι θέλουν να αναδιοργανώσουν την πόλη ε, την, ε, ε, κατόπιν δύο σεισμών εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε χάσει ένα μεγάλο πολιτισμό θα μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε από τους υπευθύνους να το περιλάβουν στις πολιτισμούς πολιτιστικές κληρονομιές και να μπορέσουν οι κάτοικοί του να το διατηρήσουν για το μέλλον προς όφελος ολονών μας και όχι μόνο της Κίνας. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ρέπο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, το ψήφισμα αυτό αφορά αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας. Αυτή η πόλη είναι μία από τις πλέον σημαντικές μουσουλμανικές πόλεις στην από Ανατολή. Ήταν μέρος ε, του δρόμου του μεταξύ που ένωνε την Ασία με την Ευρώπη και έχει τεράστια πολιτιστική κληρονομιά για το σύνολο του κόσμου. Ως εκ τούτου χρειάζεται να αναλάβουμε δράση η οποία θα προστατεύσει αυτήν την ε, πόλη από την καταστροφή. Υπάρχει επίσης και το ζήτημα της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς ε, και της πολιτιστικής ταυτότητας Πρέπει λοιπόν ε, να ξεβρεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για να προστατεύσουμε την πόλη αυτή και την, πολι... την πολιτική ταυτότητα αυτής. Ευχαριστώ. Τώρα ξεκινά η, κυρία, η διαδικασία Καζουδιά και πρώτα η κυρία Μακοβέ για ένα λεπτό οι μελλοντικέ ε, γενναίες εξαρτώνται από δικές μας ενέργειες σήμερα για να προστατέψουμε ιστορικούς τόπους όπου το Κασκαρ είναι ένας ε, βασικός ιστορικός πυλώνας του Ισλάμ στην ε, Ασία. Τώρα, το 2009 δημοσίευσε ένα πρόγραμμα η Κινέζικη Κυβέρνηση με στόχο να αντικαταστήσει το 85% της πόλης με σύγχρονα διαμερίσματα. Θα πρέπει να σταματήσουν οι η καταστροφή της αρχαίας πόλης του Κασκάρ θα πρέπει ολόκληρος ο δρόμος του μεταξιού να τεθεί υπό την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Καλούμε την Κομισιόν να θίξει το θέμα αυτό στις κινέζικες αρχές. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. Uh, Ευχαριστώ. Η πολιτική κληρονομιά είναι πολύ σημαντική για την προστασία τη πολιτική ταυτότητα. Αυτό είναι σημαντικό τόσο για την Ευρώπη, όσο για την Κίνα, όσο και τι υπόλοιπε περιοχέ. Από ό,τι είδαμε, η Κίνα έχει καταστρέψει πολλές περιοχές όπως το Θιβέτ και τώρα πράττει το αυτό στο Κασκάρ. Θα πρέπει λοιπόν για μια ακόμα φορά να εξηγήσουμε ποια είναι η θέση μας και να ζητήσουμε ρητά από την κινέζικη κυβέρνηση να σταματήσει την πολιτική καταστροφή του Κάσκαρ που είναι ένα αρχιτεκτόνημα το οποίο θα πρέπει να κρυθεί διατηρηταίο και να μην συνεχιστεί η ανοικοδόμηση που προβλέπεται. Επίσης η Κίνα θα πρέπει να κρυφθεί και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις μειονότητες. Εάν θέλει να την αντιμετωπίζουμε ισότιμη, χρειάζεται να δείξει σεβασμό απέναντι στις μειονότητες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ρομέδε Ρουέντα. Το λόγο το έχει, έχει ο κύριος Ρούμπι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Επίτροπε Χάν. Νομίζω ότι ο πολιτισμός και η ταυτότητα διεθνώς πρέπει να τονιστεί και ε, όπως ελέγχθη ήδη πρέπει να θεωρήσουμε πολύ σημαντικό η κληρονομιά αυτή να μην παραμείνει μόνο στην διάθεση των Ιουγούρων αλλά προς όφελος της διεθνούς κοινότητος και η Κίνα θα πρέπει να κάνει ένα βήμα για να μας προσεγγίσει διότι το ίδιο έγινε με την πόλη Βεντζού όπου μπορεί κανείς πλέον να επενδύσει κατευθείαν σε δολάρια και πιστεύω ότι και σε αυτή την περιοχή μπορούμε να πράξουμε το ίδιο, να υπάρξουν τα ίδια δικαιώματα όπως σε άλλες περιοχές της Κίνας και οι διεθνείς σχέσεις θα τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Και τώρα η κυρία εσάγια έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα βασικά δικαιώματα των μειονοτήτων στην Κίνα δεν γίνονται σεβαστά. Μιλώ φυσικά για εθνοτικές μειονότητες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αρνείται τη δυνατότητα το, στο Κάσκαρ να διεκδικήσει το καθεστώς παγκόσμιας πολιτικής, πολιτιστικής κληρονομιάς. Κλείνει τα πολιτιστικά κέντρα στο Κάσκαρ και δεν βρίσκεται το Κασκάρ στον κινέζικο κατάλογο των ε, μεγάλων ε, των ε, κτηρίων μάλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προσπαθούν να αρνηθούν αυτήν την κληρονομιά στις μελλοντικέ γενναιές, να καταστρέψουν αυτή την πόλη και βία επιτίθεται στην πολιτιστική κληρονομιά των Ιγούρων. οι Κινέζοι δηλαδή αρνούνται το γεγονός ότι, ότι οι ίδιοι είναι μια πολυπολιτιστική κοινωνία. Ευχαριστώ τη συνάδελφα Ισάγια. Ο κύριος Ζανέσκη έχει ένα διαδικαστικό. Έχετε διαδικαστικό? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο επί του θέματος αυτού. εσείς κάνατε το σήμα, το διεθνές σήμα για ε, καδιαδικαστικό. Διαφορετικά τώρα είμαστε στη διαδικασία κάτσου διάει και δεν πάει έτσι. Πρόεδρε, ο λαός των Ιγούρων πραγματικά κινδυνεύει. Αυτό ε, το ε, πρόγραμμα αστικής ανοικοδόμησης ε, θα καταστρέψει τον πολιτισμό στην περιοχή, όπως επίσης θα καταστρέψει και την αρχαία πόλη, αλλά και τον δρόμο του μεταξιού. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από το να παραβιάζουν τα δικαιώματα των μειοτήτων. Το Κασκάρι είναι ένα από τα καλύτερα αρχιτεκτονήματα της περιοχής μπορούν ε, να να ανα, μπορεί να αναπλαστεί η περιοχή, μπορεί να αναπαλαιωθούν τα κτίρια, αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται να ανοικοδομηθούν. Θα μπορούσα να ζητήσω την συμπερίληψη του πόλη του Κασκάρ ε, ως ε, πολιτιστικό μνημείο πάνω στον δρόμο για το, το του μεταξιού. Και ζητάμε από την Κίνα να σεβαστεί αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ, όλους του... Ευχαριστώ τη συνάδελφο Μπασέσχου και όλους οι οποίοι σεβάστηκαν το χρόνο και μπορώ να δώσω το λόγο ακόμη σε δύο υποψηφίους στη διαδικασία Κατσουδιάη, στην κυρία Κόρολα και στον κύριο Ζανέτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η περιοχή είναι πολύ μακρινή αλλά οι Ουγγόροι κατάφεραν να κρατήσουν επί χιλιετερίδες τις παραδόσεις τους και οι Κινέζοι τώρα προσπαθούν να ελέγξουν την περιοχή λόγω ενεργειακών σκοπιμοτήτων. Τα δικαιώματα όμως των μειοψηφιών πρέπει να διατηρηθούν και για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν παραδοσιακά οι Ουγγουροί ας υπάρξουν βελτιώσεις των υποδομών δεν πρέπει όμως να καταστρέψει 80% της παλιάς πόλης και να τοπίσει 20% του πληθυσμού. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν διότι διαφορετικά αυτός ο, εξωτικός πολιτισμός θα εξαφανιστεί. Ευχαριστώ και τελευταίο στη διαδικασία Κατσουδιάη έχει το λόγο ο κύριος Φερνάνσκι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ε, μπορούσα να με δείτε από την αρχή που σας έκανα νόημα. Στο Ευρωπαϊκό για μια ακόμα φορά συζητάμε για το ζήτημα της μειονότητας των ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι και στο παρελθόν είχαμε ψηφίσει υπέρ αυτής της μειονότητας και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, θρησκευτικέ μειονότητες που διώκονται όπως ε, και η χριστιανική μειονότητα η οποία διώκεται δεν ε, στηρίζεται διόλου από τις αρχές και η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να ε, υποστηρίξουμε όχι μόνο τις δικές μας αλλά και όλες τις μειονότητες ε, που ζουν στην Κίνα. Ευχαριστώ κύριε Τσανέσκη. Ευχαριστώ. Με τον κύριο Ζανέσκη ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the και τώρα έχει καταληκτικά τον λόγο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διατήρηση του, της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι κεντρική σημασία για την εξασφάλιση της προστασίας και της συνέχισης ε, παραδόσεων των μειονοτήτων, καθώς και του τρόπου ζωής τους. Επιπλέον, η καταστροφή σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς ε, μπορεί να αποτελέσει σοβαρό χτύπημα, όχι μόνο για την ίδια την κληρονομιά και την αρχαιολογική κληρονομιά της εν λόγω μειονότητας, αλλά και για την πολιτιστική κληρονομιά εν γέννη. Ε, αυτό το, την οπτική γωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ανάπτυξη της ε, αυτόνομης περιοχής αυτής της ε, περιοχής της Κίνας. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των μειονότητας των Ουιγούρων στην πολιτιστική κληρονομιά ε, της Κίνας. Το Κάσγαρ είναι μια περιοχή αρχαία. Το 2009 δηλώθηκε ότι η αποκατάσταση του Κασκάρ είναι απαραίτητη για να προστατευτεί η πόλη από σεισμούς ή πυρκαγιές. Αυτό είναι ένας ε, σωστός στόχος. Η κοινωνία των πολιτών στην Κίνα αλλά και διεθνώς έχει εκφράσει μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται διότι φοβούνται ότι μέχρι και το 85% της παλιάς πόλης μπορεί να ε, καταστραφεί πολλά σημαντικά κτίρια όπως το, το θρησκευτικό σχολείο ε, Σαν Λίκ φαίνεται ότι ήδη έχει καταστραφεί και 200.000 άνθρωποι να μεταφερθούν από τα σπίτια τους και φαίνεται να μην υπήρξε καθόλου διαβούλευση με τους ε, άμεσα ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν φόβοι πως η καταστροφή δομών που έχουν αποτελέσει τη βάση της ε, κουλτούρας των Ουιγούρων εδώ και εκατοντάδες χρόνια μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο για την διατήρηση της μειονότητας τα επόμενα χρόνια. Είναι επίσης λυπηρό που η Κίνα δεν πρότεινε το Κάσκαρ ως ε, χώρο πολιτιστικ, παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς παρά τη μοναδικότητά του, γιατί έτσι η UNESCO θα μπορούσε να έχει συμμετέσει στη διαδικασία της αποκατάστασης ε, της πόλης. Ε, πάντως η UNESCO ούτως ή άλλως έχει κάνει διαβήματα προς τις κινέζικες αρχές σε σχέση με τον αντίκτυπο της ανάπτυξης της παραδοσιακής κληρονομιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς του Κασγκάρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες και καλεί τις κινέζικες αρχές να συνεργαστούν με την UNESCO ώστε να εξασφαλίσουν ότι Οποιαδήποτε εξέλιξη και ανάπτυξη του Κάσκερ θα ακολουθήσει διεθνεί προδιαγραφές. Επίσης καλούμε τις ε, κινέζικες αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι κάτοικοι του Κάσκερ θα συμμετέχουν σε διαβούλευση για το μέλλον της πόλης και ότι οι υπόψει θα ληφθούν υπόψη από τι αρχέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Χάν. Κατόπιν αυτού υπάρχουν έξι ψηφίσματα τα οποία έχουν υποβληθεί. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και αρχίζει η ψηφοφορία. Καταρχήν για το Πακιστάν.